Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι συνεργάστηκαν για αυτή την έκθεση, ιδίως τους και για τη δική του συμβολή, για το αυτοσιωμένο τους έργο για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε τροπολογίες συμβασμού. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον καθηγητή Κράσνοντέσκι για τη δική του γνωμοδότηση από την πλευρά της Επιτροπής Πολιτισμού και όλους τους συναδέλφους οι οποίοι υπέβαλαν τροπολογίες. Τα σχόλιά σας πράγματι βελτίωσαν την έκθεση αυτή και την έκαναν πληρέστερη. Η έκθεση για την απόκτηση δεξιοτήτων ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει καλύτερη προετοιμασία των ε, αποφύτων του σχολικού συστήματος ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες της εργασιακής αγοράς. Χρειαζόμαστε μια πραγματική εταιρική σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών και καταρτιστών και των επιχειρήσεων. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε την νεότητα σε όλες αυτές τις δράσεις που θα βελτιώσουν την κατάστασή τους στην αγορά εργασίας. Θέλουμε να εστιάσουμε περισσότερο και στο ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές στην διαδικασία δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης και στην ανάπτυξη ικανοτήτων, ιδίως όταν πρόκειται για δεξιότητες οι οποίες σχετίζονται με το πνεύμα του επιχειρήν. Η έκθεσή μου επίσης εστιάζει στις λεγόμενες κέρυες δεξιότητες, που περιλαμβάνουν και τις δεξιότητες που έχουν να κάνουν με τις νέες τεχνολογίες και το πόσο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να συνδέσουμε την ακαδημαϊκή παιδεία με διαδικασίες μαθητείας στην πραγματική οικονομία. Μας ε, ενδιαφέρει λοιπόν η παιδεία να έχει πιο ευέλικτο χαρακτήρα και να προσαρμόζεται περισσότερο. Βασιζόμαστε στην διαβίω εκπαίδευση και την άρση των εμποδίων για την κατάρτιση και την επανακατάρτιση. Θέλουμε λοιπόν οι δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν <clears throat> για την ε, περαιτέρω παιδεία στο χώρο εργασίας να βελτιωθεί γιατί προς το παρόν είναι ανεπαρκής. Είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε και τις ανάγκες των ομάδων που είναι μειονεκτικές. Για τα παιδιά από οικογένειες μεταναστών και επίσης για νέους οι οποίοι έχουν μειονεκ... Ε, έχουν αναπηρίαση άλλα μειονεκτήματα. Είναι απαραίτητο να εστιάσουμε σε αυτές τις ομάδες και να βελτιώσουμε τις ικανότητές τους σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες. Στην έκθεσή μου εγώ δίνω μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι τα ταλέντα, οι αξίες, οι προτεραιότητες των νέων που έχουν μεγαλώσουν την εποχή <clears throat> ταχείας και ραγδαίας τεχνολογικής ε, πρόοδου είναι πολύ διαφορετικές από αυτές των προηγουμένων γενναίων. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτό το δυναμικό για την νεότητά μας που δεν έχει γίνει δεν έχει χρησιμοποιηθεί πλήρω γιατί δεν έχει κατανοηθεί. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να ενθαρρύνουμε και να επενδύσουμε σε προγράμματα τα οποία θα κάνουν πιο εύκολα τους, ε, στους εργοδότες και στους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιήσουν για να κατανοήσουν καλύτερα τις δυνατότητες των νέων μας. Είμαι πεπισμένος ότι αύριο θα ψηφίσουμε, που θα ψηφίσουμε αυτή την έκθεση, θα στεφθεί υπό επιτυχία στο κοινό μας έργο και θα οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικές δράσεις που θα υποστηρίξουν τους νέους μας στην αγορά εργασίας. Ελπίζω ότι τα συμπεράσματα αυτής της έκθεσης θα είναι και έμπνευση για περαιτέρω εργασίες. Με τα πάρα πολύ ψηλά επίπεδα ανεργία στην Ευρώπη έχουμε ένα τρομερό κίνδυνο για το κοινωνικό και οικονομικό μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όποτε μιλάμε για νέους και απασχόληση, λέμε οι νέοι θα πρέπει να κάνουν αυτό, οι νέοι θα πρέπει να κάνουν το άλλο. Οι νέοι δεν χρειάζονται συμβουλές από μας Αυτό που χρειάζονται είναι στήριξη και αποφασιστικότητα εκ μέρους μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν είναι αρκετά μεγάλη για το, τα ταλέντα τους και το Εράσμος θα πρέπει να ανοίξει σε όλο τον κόσμο. Θα πρέπει να γίνει παγκόσμιο πρόγραμμα. Έτσι οι Βούλγαροι, οι Κροάτες, οι Γερμανοί θα γίνουν ανταγωνιστικοί έναντι των Ρώσων, των Κινέζων και των Αμερικανών. Οι νέοι θα πρέπει να ε, μπορούν να ε, να μείνουν μακριά από τα γραφεία έβρεση εργασία. Κάποιοι λένε ότι η γενιά αυτή είναι μια χαμένη γενιά. Όχι, δεν είναι σωστό. Ε, οι νέοι είναι η ραχοκοκαλιά του μέλλοντος, όχι η ουρά του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η ενεργεία των ε, νέων στην ε, Ευρώπη είναι μια βόμβα η οποία μπορεί να καταστρέψει το μέλλον μας. Είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστεί. Δεν έχουμε δικαιολογία ε, όταν θυσιάζουμε τους νέους. Στη δική μου εκλογή περιφέρεια έχουμε πολύ ψηλά ε, ποσοστά νεανικής ανεργίας ε, και γι' αυτό προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε δυνατότητες και κονδύλια. Ε, υπάρχει δυνατότητα να καταπολεμηθεί η ανεργία δημιουργώντας ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους και σίγουρα βέβαια είναι σημαντική η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η μαθητεία. Μην δαιμονοποιούμε τους νέους. είναι η έλλειψη αξιοπρεπών θέσεων εργασίας που πρέπει να μας απασχολήσει. πολλοί άνθρωποι ε, πολλοί νέοι άνθρωποι ε, έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες αλλά πρέπει να σπάσουν αυτό το φαύλο κύκλο που υπάρχει ε, χαμηλή αμοιβή, εκμετάλλευση δημιουργούν μια νέα ορολογιακή βόμβα θα πρέπει να την απενεργοποιήσουμε για να ενεργοποιήσουμε τους νέους στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς κύριε πρόεδρε από τη στιγμή που η τρόικα άρχισε να εφαρμόζει τις μνημονιακές πολιτικές το ποσοστό της συνολικής ανεργίας αλλά και της ανεργίας των νέων στην ελλάδα κατέστη το υψηλότερο στην ευρωπαϊκή ένωση. επίσης πρόσφατες εκθέσεις του οσα τοποθετούν την ελλάδα στην πρώτη θέση παγκοσμίω σε ποσοστό ανέργων πτυχιούχων με 19,4% τέσσερα και ενώ η χώρα βρίσκεται στη λίστα των δέκα εξυπνότερων του κόσμου που διαμορφώνεται στη βάση του αριθμού πτυχιούχων στου τομεί των τεχνολογιών και τη επιστήμης. Όπω είναι αναμενόμενο η κατάσταση αυτή οθεί χιλιάδε νέου στην αναζήτηση εργασία στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στι χώρε δανειστέ όπω τη γερμανία που βρίσκουν ένα φτηνό υψηλά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό χωρί να έχουν ξοδέψει ούτε ευρώ για την εκπαίδευσή του. τα πρωτοφανή αυτά φαινόμενα απεικιοκρατική αφέμαξη εγκεφάλων brain drain θα καταπολεμηθούν μονάχα με την κατάργηση των μνημονίων που θέτουν τις οικονομίες της ευρωπαϊκής περιφέρειας σε καθεστώς ομοιρίας από τους δανειστές απορροφώντας την κύρια πηγή πλούτου τους δηλαδή τους ανθρώπους τους. ευχαριστώ. Θέλω να τονίσω την ανάγκη συνέργειας μεταξύ βιομηχανίας και εκπαιδευτικού συστήματος. Πρέπει να υπάρχει μια εταιρική σχέση εδώ. Ειδικότερα θέλω να τονίσω το ρόλο του τουρισμού, γιατί οι νέοι ακόμη και αν δεν έχουν τις ε, ειδικέ δεξιότητες μπορούν εκεί να βρουν δουλειά. Ζήτησα το λόγο για να τονίσω δύο πράγματα. Πρώτον, την αυταπασχόληση των νέων. Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο για να δώσουμε κίνητρα στους νέους, ώστε να αρχίσουν μια δική τους δουλειά. Δεύτερον, η μικροχρηματοδότηση. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν δυνατότητες ε, μικροχρηματοδότησης. Αυτά τα δύο πρέπει να ε, εισαγάγουμε στην έκθεση για να τη βελτιώσουμε. Ευχαριστώ, κύριο Φεραίρα. Είναι προφανές ε, ότι η ανεργία στο 30% <laughs> δεν δημιουργεί ελπίδες για τους νέους. Οι πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ε, στις χώρες ε, που έχουν μνημόνιο, έχει καταδικάσει τους νέους ε, στην επισφάλεια, στην ανεργία και στη μετανάστευση. Η, παιδεία έχει γίνει, ε, έχει εμπορικοποιηθεί ε, και ε, η, η εκπαίδευση προσανατολίζεται μόνο στις ανάγκες της αγοράς. Αυτό δημιουργεί δραματική κατάσταση σε, εκατομμύρια νέους. Δεν είναι δυνατόν να πουλάμε ψεύτικες λύσεις όπως η επιχειρηματικότητα που είναι μια επινόηση του νεοφιλελευθερισμού. Η λύση είναι να σταματήσουμε αυτές τις πολιτικές και να απομακρυνθούμε από αυτούς που τις προωθούν. Ευχαριστώ. Σόλτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο δημιουργεί προβλήματα στην Ευρώπη και αυτό ισχύει και πριν από την κρίση και φυσικά συνέχισε και μετά την κρίση. και στην προηγούμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μίλησαμε για τις δυσκολίες να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία των νέων. Τα στοιχεία είναι εύγλωτα. Είναι πάρα πολλοί οι νέοι που είναι άνεργοι σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ό,τι μπορεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιορίζει κονδύλια για αυτή την κατεύθυνση, αλλά αυτό δεν είναι επαρκές. Πρέπει να προσδιορίσουμε κονδύλια τα οποία θα οδηγήσουν σε θέσεις μόνιμες και υψηλής ποιότητας. Δεν είναι αρκετοί οι νέοι οι οποίοι εμπλέκονται στην αντιμετώπιση <clears throat> του προβλήματος αυτού και στη διαμόρφωση των προγραμμάτων και όπως είπαμε πολλοί συνάδελφοι, σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές χώρες έχουμε θέσεις οι οποίες είναι μονάχα επισφαλείς φτάνουν πολλές φορές το 40 ή το 60% των νέων θέσεων εργασίας. Αυτό φέρνει τους εργαζόμενους και τους νέους σε μόνιμη αβεβαιότητα, δεν μπορούν να δημιουργήσουν οικογένειες. Ευχαριστώ. Κύριος Μπάτεν. Σας ευχαριστώ. Η ανεργία των νέων στην Ευρώπη έχει φτάσει σκανδαλώδη επίπεδα και υπάρχουν δύο κύριες αιτίε για αυτό το φαινόμενο. Αυτό είναι το ενιαίο νόμισμα και το άλλο η υπερβολική ρύθμιση των επιχειρήσεων. Η Βρετανία είναι στο ευρώ και έχουμε όμως να αντιμετωπίσουμε την υπερβολική ρύθμιση. Δεν είμαστε στο ευρώ, αλλά έχουμε την υπερβολική νομοθεσία. Έχουμε πάρα πολλούς μετανάστες εργαζόμενους που φεύγουν από τις καταραίουσες οικονομίες τους. Είχα μία <clears throat> συζήτηση με ένα νέο Βρετανό στο Λονδίνο, ο οποίος δούλευε ευκαιριακά στον ε, ε, το κατασκευαστικό του είπαν ότι θα δεχτείς μια μία στον αποδοχό σου ή θα σε αντικαταστήσουμε με κάποιον από την Ανατολική Ευρώπη. Δεν μπορούν λοιπόν να ανταγωνιστούν με τη φτωχή, φθηνή εργασία που θα δουλέψουν για ψίχουλα. Οι Βασίλειο πρέπει να υποστηρίξουν τον μέλλον τους με το να υποστηρίξουν στο επόμενο δημοψήφισμα την έξοδο των Βρετανών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Πλούρα για την έκθεση. Όπως ακούσαμε η νεανική ανεργία είναι προφανώς από τις μεγαλύτερες σημερινές προκλήσεις στην Ευρώπη και για να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά πρέπει να βελτιωθούμε ε, στην προσπάθεια ε, προσφοράς και ζήτησης, προσφοράς ειδικοτήτων των νέων και ανάγκες ε, της βιομηχανίας. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία μεταξύ τοπικών αρχών, επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ούτως ώστε να καλύπτεται η ανάγκη της αγοράς. Η μαθητεία είναι πολύ σημαντική. Η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση είναι σημαντική εδώ. Ε, θα πρέπει να περάσουμε ομαλά, να περνούν ομαλά από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Και ε, υπάρχουν και ειδικότητε που ε, αποκτώνται με μη τυπικό τρόπο. Αυτές θα πρέπει να αναγνωρίζονται καλύτερα μέσα από τον εθελοντισμό ή οτιδήποτε. Ε, όλα αυτά είναι προτεραιότητες. θα, την Οκτώβριο θα υποβάλλουμε έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος και πόσο τα κράτη-μέλη ε, έχουν καλύψει ε, τις ανάγκες που υπάρχουν σε σχέση με ένα πλαίσιο ε, ποιοτικό για τις ειδικότητε. Είναι σημαντικό και το θέμα της προχρηματοδότησης από 15% στα 30% η αύξηση έγινε δεκτή από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο οπότε έχουμε μία προκαταβολή περίπου 1 δις ευρώ προς τα κράτη-μέλη για το σκοπό αυτό. Ε, άλλα προβλήματα που αναφέρονται στην έκθεση. Ε, η ανάγκη προώθησης ίσων ευχαιριών, επιχειρηματικότητας, ευελιξίας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Όλα αυτά είναι θέματα που απασχολούν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάρχει πρόοδος στις εργασίες εδώ. Ε, θέσαμε προτεραιότητε πέρσι για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και το πλαίσιο εκπαίδευση κατάρτιση 2020. Το Νοέμβριο η Κομισιόν άρχισε μια πρωτοβουλία συνεργασίας με τις επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερομένους για ένα σύμφωνο για την νεολαία. Με τη βοήθεια των επιχειρήσεων αυτό το σύμφωνο ε, θα εξασφαλίσει εταιρικές σχέσεις 10.000 ε, ε, και 100.000 νέες ευκαιρίες για τους νέους. Η καλή είσοδο συνεργασία θα εξασφαλίζεται όπως και η καλή ε, απόδοση στην εργασία. Ε, θα βοηθήσουν ε, εδώ και οι θέσεις μαθητείας που αυξήθηκαν σε 140.000 Υπάρχει και με ένα νέο θεματολόγιο για τις νέες ειδικότητες δεξιότητες, πάνω σε αυτό εργαζόμεθα. Θέλουμε το θεματολόγιο αυτό να συμπεριλαμβάνει απτές δράσεις για να βελτιώσει τη σημασία εκπαίδευση και κατάρτιση σε ολόκληρη την Ευρώπη και η έκθεσή σας θα είναι μεγάλη βοήθεια για να ε, διαμορφώσουμε τη δουλειά μας σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. <clears throat> Με την παρέμβαση σας κλείνει η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο.